Δεν έχω λάβει αιτήματα για την τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Ούτε για αύριο. Για την Τετάρτη. Η ομάδα του ECR ζήτησε η δήλωση του Προέδρου και του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το άρθρο 50 και την εφαρμογή του κράτου από το των μελών να γίνει το πρωί και να συνοδευτεί από ψήφισμα. Ο κύριο Λόνεν ζήτησε το λόγο για να μιλήσει για το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λοιπόν τι πιο σημαντικέ διαπραγματεύσει μπροστά μα που έχει κάνει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιστορία τη, για το Brexit. Και στο Κοινοβούλιο λοιπόν αυτό ψάχνουμε να βρούμε ευρείε πλειοψηφίε στι περιπτώσει αυτέ μέσα και πάνω από όλε τι ομάδε, προκειμένου να έχουμε ισχυρή τοποθέτηση στι διαπραγματεύσει ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώπιον του Συμβουλίου. Και τι βλέπουμε λοιπόν τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ξαφνικά ο κ. Φερχόφστατ ε, διορίστηκε υπεύθυνο για τον συντονισμό των διαπραγματεύσεων αυτών ε, από πλευρά του Κοινοβουλίου, από τη διάσκεψη των Προέδρων, χωρί συζήτηση, χωρί να το ψηφίσουμε. Αυτό με εκπλήσει και συχνά μιλάμε για δημοκρατικό έλλειμμα. Αλλά όταν ε, βλέπουμε αρχηγό τέτοιων των ομάδων να αναλαμβάνει τέτοια καθήκοντα, θα ήθελα να ζητήσω να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη για να το συζητήσουμε και φαντάζομαι ότι ο κ. Περχόφστα θα ήταν υπέρ να συζητηθεί το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρα. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ποιος θα ήθελε να μιλήσει υπέρ του αιτήματο αυτού. Υπέρ. Ε, θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τη σύσταση του ECR. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η διάσκεψη των Προέδρων επέλεξε τον κύριο Φερχόφστατ ο οποίος θα διαπραγματευτεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit. Είμαι στο Κοινοβούλιο εδώ και έξι χρόνια και ακούω τα αφλήνα θύματα του κυρίου Φερχόφστατ και την τελευταία φορά είπα ότι θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι έτσι ώστε να φτάσουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι ότι για κανέναν δεν ωφελεί ο διορισμός του κυρίου Φερχόστατ ούτε για τους Γάλλους αγρότες, ούτε για την αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα να υποστηρίξετε έναν πιο ουδέτερο υποψήφιο. Το αίτημα είναι προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις για την ε, θέση σε ισχύ του άρθρο 50 μετά από αίτημα του κράτους μέλους. Ε, θα ήταν καλό να ε, ενεργοποιηθεί το άρθρο 50 φυσικά, αλλά δυστυχώς δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω γιατί και πώς λοιπόν ε, καταφέρετε αυτό το αίτημα. Ο κύριος Γκονσάλες Πόνς όμως θέλει να πάρει το λόγο να μιλήσει κατά του αιτήματος αυτού. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω αν η συζήτηση για την εφαρμογή του άρθρου 50 είναι το θέμα μας ή ο διορισμός του κ. Φερχόφστατ. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω το να ζητείτε μια συζήτηση για ένα άρθρο το οποίο ακόμα κανείς δεν έχει ζητήσει να εφαρμοστεί. Ε, τρίτον, δεν έχει νόημα η Βρετανική κυβέρνηση να έχει ζητήσει δύο χρόνια να σκεφτεί αν θα ζητήσει την εφαρμογή του άρθρου 50 και εμείς να πρέπει σε δύο μέρες να λύσουμε όλο αυτό το θέμα. Ε, η συζήτηση πρέπει να είναι τόσο σοβαρή όσο και η κατάσταση. Τέταρτον, ε, είναι τελείως επιδερμικό ένα τέτοιο σημαντικό θέμα να ζητείτε να λυθεί ε, εντάχει, πρόχειρα και χωρίς συζήτηση. Ε, προφανώς δεν βρίσκονται όσοι το ζητούν στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχει κοινοβουλευτική διαδικασία και όταν φτάσει εκείνη η στιγμή θα ενεργοποιηθεί και το Κοινοβούλιο θα το συζητήσει. Να σας πω επίσης ότι θα πρέπει να οργανωθείτε λίγο καλύτερα, διότι ενώ εσείς ζητάτε το Κοινοβούλιο να συζητήσει το άρθρο 50, που κανείς δεν έχει ζητήσει την εφαρμογή του, κάπου αλλού θα συζητείτε ο διορισμός του καινούριου Βρετανού Επιτρόπου που θέλει να γίνει μέλος θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή το ένα ή το άλλο. Μην είστε αντιφατικοί μεταξύ σας. Για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Ευχαριστώ. Ονομαστική κλίση λοιπόν είναι το έτοιμο αυτό, όπως έχει και ζητηθεί. Παρακαλώ λοιπόν, χρησιμοποιήστε τις κάρτες σας και να ψηφίσουμε. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ψηφίσατε παρακαλώ όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται το αίτημα. Και για την ε, Τετάρτη, οι Σοσιαλιστές και οι Δημοκράτες συζητούν οι δηλώσεις ε, του Συμβουλίου και της ε, Επιτροπής για την απαραίτητη ενδεχόμενη επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης να μπει το πρώτο θέμα, ως πρώτο θέμα μετά το μεσημερινό διάλειμμα και να ακολουθήσει ψήφισμα. και στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να παραταθεί η σύνοδο μέχρι τις 11 το βράδυ. Κύριος Πετέλα, υπέρ. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της ε, υποαπασχόλησης. Μιλάμε για την Caterpillar, ε, στο Βέλγιο και για την Άλστον στη Γαλλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό μέσα στα πλαίσια της βιομηχανικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Και θα πρέπει η Ευρώπη να καταβάλει κάθε προσπάθεια να αποσοβήσει τις ε, καταστροφικές αυτές καταστάσεις. Υπέρ του αιτήματος αυτό το λέγω έχει ο κύριος ε, Στάνης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Νομίζω ότι το αίτημα του Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για ε, του κυρίου Πιτέλα είναι πολύ δικαιολογημένο γιατί αυτά που συμβαίνουν ε, στη Βαλονία, στο Σαλερουά, στην Κιωσελή είναι ένα μαζικό κίνημα ανεργίας. 2.200 θέσει εργασία που είναι στον αέρα και πάρα πολλέ άλλε μαζί του ε, σε ό,τι αφορά την, το εργοστάσιο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν να γνωρίζουμε πιο πολλά Ξέρουμε ότι η Caterpillar είναι μια εταιρεία η οποία στα χαρτιά έχει κέρδος, που ε, δίδει όλο και μεγαλύτερα μερίσματα στους μετόχους τους και παρά όλα αυτά κρατά σε τέτοια κατάσταση τους ε, υπαλλήλου τη. Νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε πάσα υποστήριξη προς την κατεύθυνση αυτή. Σας ευχαριστώ. Κατά του αιτήματος, το λόγο θα πάρει ο κ. Κάζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ιδιαίτερα ατυχής κατάσταση. Είχαμε συμφωνήσει να γίνει συζήτηση. Αλλά μέχρι ότι έχουμε επαρκείς πληροφορίες, γιατί δεν τις έχουμε επί του παρόντος, νομίζω ότι αυτό το ψήφισμα δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να γίνει συζήτηση και έχουμε μια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν στην περίπτωση της ε, Caterpillar και νομίζω ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Όμως αντιτιθέμεθα σε αυτό το ψήφισμα και είμαστε κατά τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και θα ψηφίσουμε. Α, κύριος Μαριάς, έχει ζητήσει διαδικαστικό για διαδικαστικό το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, απλά θέλω να δηλώσω ότι στην προηγούμενη ψηφοφορία ψήφισαν την, προ... πρόταση του ECR, αλλά δεν δουλεύει το σύστημα δεν καταγράφηκε. παρακαλώ να το λάβετε υπόψη. εγώ ψήφισα αλλά εδώ η κάρτα μου δεν δούλευε με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί η θετική ψήφο υπέρ του ecr στην προηγούμενη ψηφοφορία. Μάλιστα, θα το συμπεριλάβουμε στα πρακτικά. Και να παρακαλέσουμε και έναν τεχνικό να κοιτάξει το μηχάνημα. Τώρα, να ψηφίσουμε το αίτημα του κ. Πιτέλα, παρακαλώ. Ποιο είναι υπέρ του αιτήματο Να σηκώσει το χέρι παρακαλώ. Ο κύριο Βέμπερ. Συγγνώμη που σα διακόπτω και πάλι μετά το ψήφισμα. Θα θέλαμε μάλλον να ψηφίσουμε ξεχωριστά το ψήφισμα και τη συζήτηση. Εμεί είμαστε υπέρ τη συζήτηση αλλά κατά το ψηφίσμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρο. Καταρχά το αίτημα του κυρίου Πιτέλα το οποίο είναι η συζήτηση τώρα και το ψήφισμα τον Οκτώβριο. Ποιος είναι υπέρ του αιτήματο αυτού. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας υπέρ του αιτήματο του κυρίου Πιτέλα. Τώρα συζήτηση τον Οκτώβριο ψήφισμα. Εάν το παρακαλώ όλοι, συνάδελφοι, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και έτσι λοιπόν θα παραταθεί η συνεδρίαση τη Ολομέλη μέχρι τα μεσάνυχτα. Με ενημέρωσαν επίση οι συνάδελφοι ότι για την τρέχουσα συνεδρίαση, το, μάλλον για τη συνεδρίαση αυτή, το Συμβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο παρόν για την Τετάρτη το απόγευμα. Εγώ θα σας παρακαλούσα να ασκούσαμε πίεση. Με τόσου προέδρου και τόσου υπουργού και τόσου εκπροσώπου τη κυβέρνηση, κάποιο δεν μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να έρθει να παρευρεθεί. Η ΓΚΟΕ, η ομάδα τη Γκουε για την πέμπτη ζητά την προφορικό ερώτημα τη Επιτροπή Απασχόλησης για τις αελάχιστους κατά τους μισθού, να πάει από την πέμπτη το απόγευμα στην πέμπτη το πρωί και να το κοιτάξουμε ε, κατευθείαν στην αρχή. Αυτό λοιπόν θα σημαίνει που σας είπα ότι θα ξεκινούσε η συνεδρία στις 8 η ώρα το πρωί. Το λόγο λοιπόν θα πάρει ο κύριος Λόπες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Την Πέμπτη το πρωί έχει προβλεθεί μια σημαντική συζήτηση για δύο έγγραφα της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, βρισκόμαστε σε μια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 125 ε, εκατομμύρια φτωχούς, 30 εκατομμύρια ανέργους. Δεν δικαιολογείται λοιπόν από αυτή τη συζήτηση να διαχωριστεί το θέμα ε, της προφορικής ερώτησης η οποία έχει τοποθετηθεί την πέμπτη το απόγευμα. Υπ' αυτήν την έννοια ζητούμε το θέμα της προφορικής ερώτησης να προστεθεί στα δύο έγγραφα τα οποία θα συζητηθούν το πρωί για θέματα απασχόλησης και το απόγευμα να συζητηθεί η προφορική ερώτηση τη Επιτροπή Πολιτισμού. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο υπέρ του αιτήματο του, του κυρίου Λόπε. Ο κ. Ηλικιώτη. Ναι, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Εξάλλου την Πέμπτη το πρωί έχουμε και άλλα θέματα τη Επιτροπή Απασχόληση. Ιδιαίτερα το θέμα του κατώτατου μισού στη σημερινή Ευρώπη που υπάρχει οικονομική κρίση ε, και εκατομμύρια εργαζόμενοι βρίσκονται σε δύσκολε συνθήκε νομίζω πρέπει να είναι σε μια περίοδο που θα μπορεί να είναι ε, περισσότεροι παρόντε στην αίθουσα παρά την πέμπτη το απόγευμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατανοώ ότι το θέμα είναι ύψης της σημασίας, όμως έχουμε πολύ σημαντικές εκθέσεις, πολύ πιο σημαντικές το πρωί. Γι' αυτό δεν συμφωνούμε να περιοριστεί η συζήτηση του πρωινού ή να απαλληφθούν ορισμένα θέματα. Μην ξεχνάμε ότι και την Πέμπτη το απόγευμα πρέπει να είμαστε παρόντες. Όποιος είναι υπέρ λοιπόν του αιτήματος του κ. Λόπες παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρα στην ιδρία σας. Πέρα στις ε, ψηφορές, συγγνώμη. Έγκριση του αιτήματος. Άρα λοιπόν την πέμπτη θα ξεκινήσουμε στις 8 το πρωί. Και θα αλλάξει ούτω η ημερήσια διατάξη. Η έκθεση για τα κατώτατου μισθού θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί την ε, Πέμπτη και η προφορική ερώτηση της Επιτροπής θα μπει το απόγευμα της Πέμπτης. Δεν έχω λάβει άλλα αιτήματα για τροποποίηση της ημερήσιας διαταξής. Ο κ. Ομπερμάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι έχουμε μια πολύ σημαντική Ευρωπαϊκή ημέρα, μια Ευρωπαϊκή ημέρα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, ε, γιατί σήμερα πριν από το ε, τόσα χρόνια απελευθερώθηκε η πόλη της Βιέννης ε, από τους Πολωνούς από τους Τούρκους. Ε, και έτσι λοιπόν τους έσωσαν από τον εξισλαμισμό, τον εξισλαμισμό της Βιέννης. Βλέπουμε λοιπόν ότι τι συμβαίνει επί χρόνια στην Ευρώπη. Και θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω και να τιμήσω τους ε, γενναίους Ευρωπαίους και να αναγνωρίσω το έργο τους στον αναπαλευθέρωση της Βιέννης. Δεν ξέρω βέβαια τι έχει να κάνει αυτό με την ορίσια διάταξη, λέει ο Πρόεδρος. Μα την ξέρετε νομίζω τον κανονισμό. Μην υποκρίνεστε ότι δεν ξέρετε ότι κάνετε κατάχρηση για σκοπούς προπαγάνδας. Και τώρα να περάσουμε στη συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Λάγεν. προς τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας. Το λόγο λοιπόν έχει ο κύριος Λάγκεν, ο εισηγητής. Να ξεκινήσω. Μισό λεπτό.